So, dear colleagues... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καλωσορίζω και πάλι την δεύτερη ημέρα της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ειδικών που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ το πόσο σημαντικό θεωρούμε το ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. για την σημερινή συνεδρίαση. Όπως ξέρετε έχουμε θεματικές ε, συνεδριάσεις. Εδώ είμαστε στην ΕΚΟΝ 1 και έχει μοιραστεί σε δύο τμήματα η συνεδρίαση. Η πρώτη αφορά τα έγγραφα του Παναμά και το Bahamas Leaks ε, και τις σχετικές αποκαλύψεις και το τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε και το δεύτερο αφορό αφορά την Τραπεζική Ένωση, την Ένωση των Χρηματαγορών και την Ένωση για τις ε, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και δεδομένου του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων μάλλον δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Αλλά προσπαθήσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσο δυνατόν περισσότερους συναδέλφους ε, και προτεραιότητα θα δοθεί στο να ε, μπορέσουν να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Οπότε, κάθε βουλή θα έχει δύο λεπτά για να μιλήσει. Θα ακούσουμε 20-25 παρεμβάσεις. Άρα βεβαίως εξαρτάται και από τα αιτήματα που θα έχουμε. Να σας ενημερώσω πως υπάρχουν κάρτες ε, τις οποίες θα συμπληρώνουν οι βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές που θέλουν να μιλήσουν και θα τα δώσουν στους κλητήρες για τη συζήτηση για τα έγγραφα του Παναμά είναι το ροζ έγγραφο, δώστε το στους κλητήρες, συμπληρώστε το και δώστε το. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο για μια εισαγωγική δήλωση στον συνάδελφο Βέρνερ Λάγκεν, ο οποίος είναι πρόεδρος της ειδική Εξεταστικής Επιτροπής στο ξέπλυμα χρήματος φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ναι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα ήθελα να τα πω στα γερμανικά. Σας ε, καλωσορίζω εδώ σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, θα γίνει μια ειδική ακρόση με τέσσερις ειδικού. Ο Μαρκ Πίτ, ο καθηγητής Μαρκ Πίτ είναι ο πρώτος, από, που ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή ε, μαζί με τον καθηγητή Στίγκλιτς. Ε, κύριε Πίτς, ε, θα μας διαφωτίσετε με την πραγματογνωμοσύνη σας. Επίσης, έχουμε τρεις σημαντικούς ε, βουλευτές από διάφορες εθνικές εξεταστικές επιτροπές, Κρότα από την Ολλανδία, πρώτα απ' όλα, Αχμετ, Αχμετ Λαουεγέ, από την Βελγική Εξεταστική Επιτροπή και Κάγετ Κράινερ αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τα Οικονομικά του Εθνικού Συμβουλίου της Αυστρίας. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλό έρισμα για τις συζητήσεις μας. Εν είδη εισαγωγής, ε, να πω κάποια πράγματα για τις εργασίες μας. Ε, το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δύο ειδικέ εξεταστικές επιτροπές συγκροτήσει, τάξη 1 και τάξη 2 ε, εξετάσαμε τα Lux Leaks και τα Tax Rulings, ε, τις ε, φορολογικές συμφωνίες που συνάπτουν τα κράτη-μέλη, που όχι μόνο στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, αλλά και προβλέπουν ε, ιδιαικούς όρους για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. και προέκυψαν δύο εκθέσεις, τις γνωρίζετε. Το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία ήταν οι βασικές χώρες που συζητήθηκαν σε αυτήν την Επιτροπή. Η Επιτροπή Πάνα, Panama Papers δηλαδή, συγκροτήθηκε μετά την ε, δημοσίευση των εγγράφων από τον Μόσακ Φονσέκα, 2,8 τεραμπάιτ, τεράστιος όγκος ε, πληροφοριών, ε, τοποθετείται σε άλλο επίπεδο η δουλειά μας, όχι μόνο για την κείμενη νομοθεσία και να αυτό επιτρέπει στρέβλωση του ανταγωνισμό, αλλά ε, ό,τι έχει σχέση με ξέπλυμα ε, χρήματος, ε, παράνομα έσοδα από διαφθορά, από εγκληματική δράση και φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή που συνδέονται με αυτά. είναι διαφορετική η προσέγγιση που ακολουθούμε λοιπόν και γι' αυτό είναι σημαντικό στα πλαίσια των εργασιών μας πρώτα απ' όλα να διαφωτίσουμε το, τα, επιστημονικά, τους, ε, τα μέλη της Επιτροπής για τα επιστημονικά στοιχεία, να εξετάσουμε τι γίνεται με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους consultants, τους ενδιάμεσους, τους δικηγόρους, τις τράπεζες που διευκόλυναν αυτή τη διαδικασία και να δούμε ποιες δυνατότητες δράσης υπάρχουν για να θεσπίσουμε διεθνή πρότυπα. Τι σημαίνει Panama ε, Papers, σκάνδαλο ε, Panama Papers είναι ένα, μια ε, Διεθνή ε, τάση να κρύβονται χρήματα, να διοχετεύονται και να κρύβονται ε, πόροι από διάφορε δραστηριότητε σε φορολογικούς παραδίσους. Ε, πρόκειται για δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρά τα ποσά, όπου σημειώνεται φοροαποφυγή και φυσικά η φορολογική δικαιοσύνη πλήττεται και δυσχεραίνεται από αυτές τις πρακτικές. το, αρχίζει από το Σεπτέμβριο του 2016 τις εργασίες μας. Ε, θα κρατήσει ε, ένα χρόνο ή κατανότα τώρα 1,5 χρόνο η Επιτροπή. Το... Στη Συνδίκη Λισαμόνας προβλέπεται ε, στο άρθρο 226 αυτή η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν διαθέτουμε καμία δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε εθνικό επίπεδο. Οπότε ελπίζουμε <laughs> ότι ε, οι προσκεκλημένοι μας από τα εθνικά κοινοβούλια θα κινηθούν. Δηλαδή δεν μπορούμε ε, να καλέσουμε κανέναν υποχρεωτικά ενώπιόν μας, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις και από το 2014 έχουμε καταθέσει πρόταση στο Συμβούλιο για να βελτιώσουμε αυτή την αρμοδιότητα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, τώρα, ε, ε την ε, μεθεπόμενη εβδομάδα θα πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο και αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη ΣΥΠΑ. Έχουμε μία σειρά από καθηγητές που ήρθαν σε δημόσιες ακροάσεις και μπορώ να σας πω ότι προθέσεις έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το ζήτημα ως προς την νομοπαρασκευαστική διαδικασία Τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, country by country reporting και επίσης ε, ενοποιημένος ε, κοινή κοινή εταιρική βάση φορολογία επιχειρήσεων, οι μονοπρόσωπε εταιρείε, την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εταιρείε γραμματοθυρίδες, που δυστυχώς όπως ξέρετε υπάρχουν και στην Ευρώπη. Έχει παγώσει αυτή η πρόταση που έχουμε καταθέσει. Ε, επίσης, tax rulings, ε, τα patent boxes ε, και σε, περίπτωση, σε δύο γνωστές περιπτώσεις, όπως ξέρετε, Apple Ιρλανδία και Amazon στο Λουξεμβούργο, ε, κρεμούν οι διαδικασίες, οι εθνικές φορολογικές αρχές ισχυρίζονται ότι μόνο το κομμάτι του τζίρου που ε, γίνεται στη, στο Λουξεμβούργο και στην Ιρλανδία θα μπορέσει να υπαχθεί σε αυτόν τον ενοποιημένο φόρο. Δηλαδή, ενώ είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ε, φορολογείται μόνο το κομμάτι αυτό του τζίρου. Και τι γίνεται, ε, μόνο το 0,5% του τζίρου της Amazon και αντίστοιχα ένα πολύ μικρό ποσοστό του τζίρου της Apple τελικά φορολογούνται στην ε, Ευρώπη. Στρέβλωση του ανταγωνισμού έγιναν οι έρευνες για την Amazon, θα ακολουθήσουν και Starbucks και άλλες εταιρείες ε, και η αρμόδια επίτροπος ε, του ανταγωνισμού αποφάσισε ότι 13 ε, δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να καταβληθούν σε φόρους στην Ιρλανδία από την Apple. Είναι, υπάρχουν κενά όμως και στην Αμερικανική νομοθεσία, λέει ο Αμερικανός νομοθέτης, πως τα κέρδη που προέρχονται από όλες περιοχές του κόσμου και μεταφέρονται υπεράκτια ή οπουδήποτε άλλο, θα πρέπει παρόλα αυτά να υπαχθούν σε αμερικανική φορολογία αν τελικά καταλογιστούν ε, στις ΗΠΑ. Ε, ένα, αν υπάρχουν 1,3 δις αποθηκευμένα σε οποιονδήποτε φορολογικό παράδεισο παραδείγματο χαρέ και τελικά έχει καταβληθεί ένας ελάχιστος φόρος παρότι στην Ιρλανδία ο τζίρος της Apple από την Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Βόρεια Αφρική ε, και την Μέση Ανατολή τελικά περνάει από την Ιρλανδία λοιπόν ε, πελώρια στρέβλωση του ανταγωνισμού και πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Σημαντική είναι η συνεργασία των εθνικών αρχών και η σύναψη διεθνών συμφωνιών. Ξέρουμε βεβαίω ότι έχουμε περιορισμένη αρμοδιότητα διότι ε, η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα Είμαστε πεπισμένοι όμως ότι ε, απαιτείται διεθνή πίεση για να ενισχύσουμε τη φορολογική δικαιοσύνη. Αυτά ήταν μια μικρή έκθεση υπεπραγμένων. Ε, το δεύτερο ήμιση του 2017 κατά πάσα πιθανότητα θα καταθέσουμε την τελική μας έκθεση από τους δύο συνεισηγητές Γέφο Κόφορτ από τους ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και Πίτερ Γέτσεκ από τους Φιλελευθέρους από τη Δανία. Ε, θα κατατεθεί λοιπόν αυτή η σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, ε, Langen. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάγκεν, λέει ο Πρόεδρος. Και ο πρώτος τώρα είναι ο καθηγητής κύριος Μαρκ Πίτ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας ε, πρόσκληση. Και έχουμε φτάσει, είπαμε, στο χειρότερο σημείο όσον αφορά ε, τα βρώμικα χρήματα. Πρόκειται για τις χώρες που δεν έχουν κάποια ε, σχετική νομοθεσία για να σταματήσει τα φαινόμενα αυτά και είπαμε ότι ένα ε, σενάριο είναι το να αγοράζουν κάποιοι δικηγόροι, κάποιες εταιρείε και έτσι να οργανώνουν τέτοια, τέτοια κεφάλαια ούτως ώστε να είναι πάρα πολύ δύσκολη συνεργασία με τις διοικητικές αρχές και ξέρετε ελβετός είμαι και ξέρω για τι πράγμα σας μιλάω όμως παρόλα αυτά εμείς ανεχόμαστε το να υπάρχουν τέτοιες χώρες που να έχουν φορολογική παράδοση να, στο ή στο στον στην, στην Καραϊβική και αλλού Οπότε ρίξτε μια ματιά τι γίνεται σε αυτά τα έγγραφα, ήδη τα είπε ο πρόεδρος και θα βρείτε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα κοκτέιλ από ε, φοροδιαφυγή, από το τραπεζικές απάτες, αλλά ακόμα και υπουργοί οι οποίοι κρύβουν λεφτά και ε, τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα από όσα θα μπορούσαν να κερδίσουν νόμιμα. Βεβαίω έχουμε και τις μαφίες, έχουμε τους ε, δουλέμπορους, ε, ακόμα και τις ε, συμμορίες που εκπορνεύουν ανηλίκους. Να, διαβάστε και το βιβλίο του Όμπερμαγερ. Και η εμπειρία μου αυτό μου είχε καταδείξει ότι τέτοιου είδους ζητήματα έχουν πάρα πολλές φορές επισημανθεί. Έχω δουλέψει στον ΟΣΑ, στα θέματα διαφθοράς και επίσης και στο πρόγραμμα για τη διατροφή του ΟΗΕ και αυτό τα έχω δει πάρα πολλές φορές, χιλιάδες φορές και όπως είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος ότι το θέμα δεν είναι μόνο ο Παναμάς, είναι απλώς ένα παράδειγμα απλώς τώρα παρεμπιπτόντω λέμε και για τον Παναμά έχω μια εικόνα και για αυτή την υπόθεση γιατί καταβάλει σημαντικές προσπάθειες τώρα η χώρα προσπαθούν να πούν αυτά που πρέπει, αλλά την ε, περασμένη εβδομάδα η έρευνα στην ε, Φωσάκα θα έπρεπε για λίγο να ανασταλεί. Γιατί ε, έτσι διέταξε ο Άριος Πάγος της χώρας. Um, Οπότε έτσι είπαμε ότι η βραζιλιάνικη εταιρεία Όλτεμπριχτ παραδέχτηκε ότι είχε πληρώσει 59 εκατομμύρια σε αυτούς που λαμβάνουν τις ε, αποφάσεις για κάποια συμβόλαια 7 δις δολαρίων και δεν έγινε τίποτα. Καμία έρευνα. Αν θέλετε, συζητήστε. Αν θέλετε ότι αυτά είναι σοβαρές κατηγορίες. Αλλά το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Όλοι είμαστε μέσα. Ε, είτε είμαστε στην πηγή του προβλήματος, είτε είτε συμβάλλουμε με κάποιο τρόπο με τους νομικούς διάβλους. Αν θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι και τολμηροί. Οπότε ήδη νομίζω ότι είμαστε σε καλή ρότα. Επανειλημμένα, ξέρετε τι γίνεται όσον αφορά ε, τους beneficial owners και τον εντοπισμό τους. Τι γίνεται πρώτα-πρώτα με τα τραπεζικά ιδρύματα και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο αν θέλετε να έχετε αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να ξέρει ε, ο καθένας σε ποιον ανήκει ο κάθε λογαριασμός, πρέπει να τα ξέρουμε και ο νομοθέτης και η ιδιοκτική αρχή. Τώρα, τι, είναι, τι λείπει από το puzzle. Λείπει σοβαρότητα στην εφαρμογή του νόμου. Να σας πω τι εννοώ. Στην πατρίδα μου, την Ελβετία, η κλασική λύση είναι Ιδίως στην Γενέβη οι δικηγόροι αγοράζουν οικοδομικές ε, εταιρείες από θηγατρική της Μόσακ Φονσέκα. Αλλά έχουμε και καταπιστεύματα, έχουμε και τους φοροτεχνικούς ε, και τους φορολογικούς συμβούλους ε, και δικηγόρους και πολλές φορές αυτά δεν είναι κλασική δικηγορική δουλειά. Πολλές φορές χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι που από εκεί που ήταν σύμβουλοι γίνονται τελικά ενεργά εμπλεκόμενοι στο χρηματοοικονομικό γίγνεσθε. Και έτσι έχουμε τώρα το, το, τον κόσμο του ξεπλήματος του χρήματος, οπότε μια νυχτή ο δικηγόρος γίνεται επομένω εκεί, εμπλεκόμενος. Άρα, αναδύεται το ερώτημα, τι να κάνουμε. Η πρώτη μου πρόταση προς εσάς θα ήταν εξετάστε προσεκτικά ποιος θεωρείται ότι έχει το προνόμιο το επαγγελματικό και της ε, επαγγελματική εμπιστοσύνη. Η με τη έτσι νομίζω ότι γίνεται. Δεν πρόκειται για δικηγόρους, δικηγόρου. Σε αυτούς δεν αρμόζει το, το προνόμιο του επαγγελματικού απορρίτου. Άρα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή στις έρευνες και στη δράση των διοικητικών αρχών. Ρίξτε τώρα μια ματιά σε αυτή την έκθεση που έγραψα με τον Τζο ε, υπάρχει αυτή η έκθεση εδώ έξω από την αίθουσα και αφορά την σκιώδη οικονομία, την παραοικονομία και λέει δύο λόγια παραπάνω αυτά που λένε τα κλασικά εγχειρίδια. Λέμε τι θα θέλαμε να ισχύσει παγκοσμίω να υπάρχουν κάποιο είδους εταιρικά μητρώα, τα οποία όμως να είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, να αναφέρονται ως εταίροι ιδρυτές εταιρείας πραγματικοί άνθρωποι. Να μην είναι κάποιος αχυράνθρωπος, να μην είναι ένας, ε, ένας κυπουρός ή η καθαρίστρια της ε, Φονσέκα που να παριστάνει την διευθύντρια. Να είναι επομένως πραγματικοί ε, ιδρυτές αυτό βέβαια είναι μεγάλο βήμα, είναι περιπλεγμένο, δύσκολο και μπλέκονται εδώ και πολλά τεχνικά ζητήματα. Θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, αλλά είμαι πεπισμένος ότι τέτοια νομοθεσία μπορεί να θεσπιστεί. Καλά, τελικά μπορεί να έχουμε όλους αυτούς τους αχυράνθρωπους στα εταιρικά μητρό, αλλά νομίζω ότι αν τελικά υπάρχει ένα μητρό εταιριών, το οποίο να έχει σημασία, να έχει ουσία, τότε μπορεί οποιοδήποτε να ελέγξει. Και αν ανακαλύψουν ότι εκεί είναι κάποιο κάποιος κάποιο δηλαδή, που δεν μπορεί, που είναι, είναι και αναλφάβητο καμιά φορά, ε, αυτό θα στριμώξει κάποιος. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι απλή πρόταση, αλλά είναι μια πρόκληση. Και νομίζω ότι ιδίω με την σημερινή συγκυρία θα πρέπει εσείς να ξεκαθαρίσετε ποια είναι η κόκκινη γραμμή όσον αφορά ε, τις ε, offshore εταιρείες. Γιατί βλέπετε ότι προσπαθούν να αντιπιτεθούν στις προσπάθειές σας οι λαϊκιστές από την μεριά του Ατλαντικού. Ευχαριστούμε καθηγητά Πίτ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που παρουσιάσατε. Όλα αυτά νομίζω αξίζει κανείς να τα λάβει υπόψη. Και θα πρέπει να θεσπίσει την νομοθεσία ούτως ώστε να προστατεύσουμε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, Ο κ. Σαντιχρόδου ο επόμενο, ο οποίο είναι ο πρόεδρο τη ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, ε, τη Ελληνική Επιτροπή για τα φορολογικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκ μέρου ε, του Ολλανδικού Κοινοβουλίου και της Αρμόδιας Επιτροπής για τα φορολογικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καλέσατε εμένα και τον συνάδελφο από τους, ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ε, τα έγγραφα του Παναμά αποκάλυψαν ε, πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στο Κοινοβουλίο της Ολλανδίας Ακούσαμε πάρα πολύ καλά την έκκληση για εξέταση της κατάστασης τον Μάιο. Η Επιτροπή Οικονομικών ε, σχημάτισε μια ομάδα εργασίας με στόχο να μάθουμε ότι μπορούμε για τις φορολογικές αυτές δομές και κατασκευές ε, και να αποφασίσουμε μετά για άλλες ε, ενέργειες. Συζητήσαμε με ειδικού, ε, παραδείγματο χάρη επιστήμονες, φορολογικούς ε, συμβούλους ε, και Ολλανδούς φορο... και υπαλλήλους της φορείας. Και καταλήξαμε τελικά ότι θα έπρεπε να κάνουμε μία μήνυ εξεταστική επιτροπή, κάτι το οποίο δεν απαιτεί μεγάλη παρασκευαστική περίοδο. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένοι να έρθουν και να καταθέσουν όρκος ε, τα άτομα τα οποία θα καλέσουμε. Κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο γίνεται στο Κογκρέσο. Πέρσι τον Οκτώβριο λοιπόν ε, εγκρίθηκε η πρόταση για εξεταστική επιτροπή και πέντε βουλευτές ε, αποτελούν αυτή την επιτροπή η οποία θα εστιάσει σε ζητήματα καταπιστευμάτων και τον ρόλο της Ολλανδίας στην διευκόλυνση των λεγόμενων εταιριών ε, γραμματοκιβωτίων. Ο βασικός στόχος είναι να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς ενεργούν και οι φορολογικοί σύμβουλοι και τα, τα πιστεύματα στην πράξη. Όπως ίσως ξέρετε η Ολλανδία είναι βασικός κόμβος των διεθνών κεφαλαιακών ροών μέσω μάλιστα συχνά εταιριών γράμματοκιβωτίων που δεν έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην Ολλανδία. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το απολύτως σύνομο. Το ερώτημα όμως είναι ε, το εάν αυτές οι δραστηριότητες ε, είναι και επιθυμητές από την οικονομική ή κοινωνική σκοπιά ή αν είναι ηθικές. Μέσω λοιπόν ε, των ερωτήσεων που κάναμε και θα κάνουμε σε αρμόδια άτομα. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποιες απαντήσεις. Θα γίνουν λοιπόν οι ακροάσεις την Άνοιξη μετά τις Ολλανδικές εκλογές και θα είναι οι ακροάσεις δημόσιες και θα μεταδίδονται από την τηλεόραση. Να αναφερθώ τώρα στο εξής. Ελπίζω ότι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα τα επόμενα χρόνια όσα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά βεβαίως η ευθύνη είναι όλων μας και των εθνικών κοινοβουλίων και του Ολλανδικού μεταξύ αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αχμέντα κατόπιν, πρόεδρος της Βελγικής Ειδικής Επιτροπής για τα Panama Papers. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ μου για την πρόσκληση. Με χαρά συμμετέχω στις εργασίες σας. Ε, θέλω να θυμίσω πω συγκρότησε μια ειδική εξεταστική επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά, το Βελγικό Κοινοβούλιο, γενικότερα όμως για τις ευρωλογικού παραδείσους και τις offshore εταιρείες. Ε, γιατί υπήρχε αυτή η ευρεία συνένεση για την ε, συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, διότι κάθε φορά που υπήρχαν ε, και αποκαλύπτωνα κύματα διαφθοράς από τον τύπο offshore leaks, lax leaks, Panama, Papers, Bahama leaks και ούτω καθεξής, Κάθε φορά ε, ε, διαπιστώναμε ότι μια σειρά από εταιρείες, μια σειρά από, ε, από του Βελγίου εμπλέκονταν σε αυτά τα σκάνδαλα. Δεν είναι μια εξεταστική επιτροπή πάντως ε, στο μέτρο που είναι περιορισμένη η αρμοδιότητα και υπάρχει ένας βασικός λόγος ε, διότι εκ παραλληλού υπάρχουν ε, δικαστικές ε, διαδικασίες ε, και φάκελοι που έχουν ανοιχθεί ενώπιον των φορολογικών αρχών και γι' αυτό δεν θέλαμε να υπάρχει ε, παρέμβαση σε αυτές τις προϊούσες διαδικασίες. Πάνω από 700, σε περιπτώσεις στα Panama Papers εξετάζονται από τις φορολογικές αρχές και συγκεκριμένα 230 φάκελοι εξετάζονται αυτή τη στιγμή από τις φορολογικές αρχές και υπάρχουν και άλλοι δικαστικοί ε, ε, φάκελοι από το ΣΕΝΤΕΦΟ είναι η αρμόδια αρχή για το δίωξη οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος. Ε, έχουμε λοιπόν αυτές τις δικογραφίες, έχουμε την αστυνομία και την Εθνική Τράπεζα που ελέγχει τους διαμεσολαβητές. Οι μεγάλες τέσσερις τράπεζες, the Big Four, πάρα πολλοί επαγγελματίες ε, εμπλέκονται. Ο δικαστής και ο ειδικό ε, εισαγγελέα, νομίζω ε, προσκλήθηκε και από την Εξεταστική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Θα γνωρίζετε τι κάνει. Προκύπτει ήδη ότι ε, χωλένουμε σε συντονισμό ανάμεσα στις συναρμόδιες αρχές για τη δίωξη οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος. Ε, βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη, η αστυνομία, η αρχή καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος, ευρώμικου χρήματος, ε, η κεντρική τράπεζα, οι φορολογικές αρχές δεν συντονίζονται επαρκώς. Δεν υπάρχει επαρκής ροή και ανταλλαγή πληροφοριών. Οπότε χρειάζεται ανάληψη μέτρων σε αυτό το τομέα. Και κάτι άλλο που επαναλαμβάνουμε διαρκώ, δεν υπάρχουν ενιαίοι κατάλογοι φορολογικών παραδείσων ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε σε επίπεδο Βελγίου. Εξαρτάται από το κεφάλαιο φορολογική απάτη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πλήρη ενιαίο κατάλογο φορολογικών παραδείσων ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το ιδιαίτερα επιζήμιο φαινόμενο. Ο Πιέρο Μοσκοβίση, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, ε, μας μίλησε στο Κοινοβούλιο και μας είπε ότι ε, προτίθεται σε αυτό το τομέα και σε ένα ε, και σε πολλούς άλλους να δραστηριοποιηθεί. Η Εθνική Τράπεζα, ενώ προβλέπεται στην αποστολή της να εντοπίζει ειδικού μηχανισμούς που διευκολύνουν τη φορολογική απάτη μέσω των τραπεζών, παρόλα αυτά διαπιστώνουμε έλλειψη αυτών αποτελεσμάτων και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, ε, θέλουμε να συγκροτηθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή για την καταπολέμηση της ε, φορολογικής απάτης. Δεν γνωρίζουν σύνορα ε, οι, όσοι διαπράττουν φορολογικές απάτες, οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφιστώ την προσοχή σας και σε κάτι άλλο χρειάζεται ενίσχυση του νομικού πλαισίου ώστε να καταστέλλονται οι facilitators, οι τράπεζες, ε, τα δικηγορικά γραφεία που χρησιμοποιούν την πραγματογνωμοσύνη για την συγκρότηση αυτών των δόλιων ε, φορολογικών μηχανισμών. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Γκουαλτιέρη. Κάι Αντιπρόεδρος Επιτροπής ε, Οικονομικών του Αυστριακού Εθνικού Συμβουλίου. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην Αυστρία είχαμε μια τράπεζα η οποία αναφερόταν στα Panama Papers, μια περιφερειακή τράπεζα που είναι ιδιοκτησία μιας περιφέρειας ε, που είναι στα σύνορα με την Ελβετία και το Λιχτενστάιν και ήταν ήδη σεσημασμένη θα λέγαμε γιατί είχε στενές σχέσεις ε, με ιδρύματα στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν και στο τοπικό κοινοβούλιο υπήρχε ήδη μια επιτροπή για να εξετάσει το ζήτημα. Η έκθεση θα δημοσιευτεί νομίζω αυτή τη βδομάδα, τα όπου να και το βασικό αποτέλεσμα ήταν πως Παρετήθηκε το ΔΣ και άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο της ε, τράπεζας και στο μέλλον θα απαγορεύονται οι σχέσεις με φορολογικούς παραδείσους και οι σχέσεις ε, με εταιρείες γραμματοκιβώτιας υπεράκτιες ε, δικαιοδοσίες από τις ε, συζητήσεις ε, στο τοπικό και στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξουν τρεις πυλώνες της πολιτικής μας. Ο πρώτος είναι η διαφάνεια με σημαντικά ζητήματα όπως ε, τα δημόσια αρχεία των εταιριών αυτών και των τελικών δικαιούχων όπως το παραδείγμα του χάρη το Μητρό των Επιχειρήσεων στη Γερμανία, όπου υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρεία, αλλά και ιδρυμάτων. Και το δεύτερο σημαντικό βήμα διαφάνειας νομίζω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εταιρείες γραμματοκιβώτια όπως λέγονται. Ο μόνος στόχος είναι η φορολογική απάτη και η αδιαφάνεια. Και πρέπει νομίζω να απαγορευτούν. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η συνεργασία μεταξύ κρατών. Μοιραζόμαστε πληροφορίες ε, ε, επί εταιριών, ε, επί φορολογικών αποφάσεων, πολλά πράγματα. Τα έχουμε ήδη δρομολογήσει μέσω οδηγιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και το ζήτημα είναι πώς θα προστατεύουμε τους πληροφοριοδότες και δεν εννοώ μόνο τους μουσιογράφους, γιατί νομίζω πως αυτό είναι σχετικά σαφές. αλλά και όσους ε, αποκαλύπτουν πληροφορίες από το εσωτερικό μιας εταιρεία. γιατί εντάξει υπάρχει βεβαίως ένα επιχειρηματικό απόρριτο, αλλά αυτό δεν μπορεί ποτέ να καλύπτει την φορολογική απάτη ή το ξέπλυμα χρήματος. Τότε, εάν κάποιος αποκαλύψει τέτοιες ε, πληροφορίες, θα πρέπει να προστατεύεται από τα κράτη μας και να μην ε, σύρεται στα δικαστήρια. Ο τρίτος ε, πυλώνας είναι η δίκαιη φορολογία, ειδικά για τις πολυεθνικές εταιρείες, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο εκθέσεις αναχώρα και άλλα πράγματα που έχουμε ήδη δρομολογήσει, αλλά επίσης νομίζω πρέπει να εναρμονίσουμε τα φορολογικά μας ε, συστήματα. Οι εταιρείε εργάζονται σε διεθνές επίπεδο και άρα χρειάζεται κάποια διεθνής ρύθμιση, διεθνής φόρη, για τις εταιρείες, δηλαδή μια κοινή φορολογική ε, βάση για τις επιχειρήσεις ή τουλάχιστον κάποιο εύρος φορολογικών συντελεστών για να μην έχουμε πάλι έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω που πάλι τελικά θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, τις φορολογικές διαφορές μεταξύ χωρών. Και πρέπει επίσης να δούμε αυτούς οι οποίοι βοηθάνε αυτή την κατάσταση και βοηθούν εταιρείε και πολύ πλούσιους ανθρώπους που προσπαθούν να μην πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί και μιλάω για τράπεζες και φορολογικούς ε, συμβούλους και νομίζω ότι πρέπει να χαράσονται τα λογιστικά πρότυπα από τους νομοθέτες ε, και όχι από κάποια ιδρύματα ε, που καθορίζουν ε, τους κανόνες. Χρειαζόμαστε λοιπόν, όπως είπαμε, τα λογιστικά πρότυπα για τη φορολογία, οπότε πρέπει να περιληφθούν στην νομοθεσία και τέλος υπάρχουν βεβαίως κάποια μέρη του κόσμου που θα συμμορφωθούν και αν δεν συμμορφωθούν κάποιος θα είναι εκτός, οπότε αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να στείλει λεφτά σε μια εταιρεία γράμματο κυβότιο, ε, τότε πρέπει να υπάρχει κάποιος δασμός ε, στα σύνορα που πρέπει να είναι περίπου το ε, ποσοστό ένα 35 με 45% ε, το ποσοστό το οποίο αναλογεί γενικά ε, στην φορολογία επί του ΑΕΠ. Ε, εντάξει, μπορεί να ακούγονται κάπω ριζοσπαστικά όλα αυτά, αλλά νομίζω είναι εύκολα. είτε κάποιο θα είναι εντός του συστήματος, είτε εκτός. Και όταν είναι εκτός, θα πληρώνει όταν βγάζει λεφτά από τη μία ζώνη στην άλλη. Όταν τα βγάζει από τον κόσμο του φωτός να πάνε στη Μόρντορ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε... Έχουμε τώρα και την ευκαιρία να συζητήσουμε τον καθηγητή Μαρκ Πίτ, ο οποίος μαζί με τον καθηγητή Ζόζεφ Στίγκλιτς ε, έκανα μία έρευνα για την σκιώδη οικονομία. Λοιπόν, 13 συνάδελφοι έχουν ζητήσει τον λόγο. Είχαμε προβλέψει να ακούσουμε τρεις ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και έναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πάμε έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 8 βουλευτές και 6 ευρωβουλευτές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα προσπαθήσω να είμαι ευέλικτος. Αν έχετε ερώτηση προς ε, κάποιον από τους τέσσερις ομιλητές, να απευθυνθείτε σε αυτόν συγκεκριμένα. Έχουμε προβλέψει δύο λεπτά για την κάθε παρέμβαση. Ξεκινάμε με τον Τζέισον Ατσουπάντη από την Μάλτα. Έχετε τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ώρα περηφάνειας γιατί η χώρα μας που αναλαμβάνει την Προεδρία. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους απεσιόδοξους, όλους τους όσους προφητεύουν το κακό και επίσης κρίμα που η Προεδρία μας σκιάζεται από το σκάνδαλο των Panama Papers και έχουμε τώρα την αμφίβολη τιμή του να είμαστε η μόνη χώρα που έχουν αποκαλυφθεί εις βάρος της κάποια τέτοια γεγονότα. Μιλάμε για χρήματα τα οποία ο εμπλεκόμενος υπουργός δεν μπορούσε ποτέ να τα έχει νόμιμα κερδίσει. Και είναι σαφές για όλους γιατί ήθελε βέβαια να έχει εταιρείε offshore. Τώρα αυτός ο υπουργό ήθελε να προεδρεύει στο Συμβούλιο Υπουργών Ενεργείας. Αυτό είναι ντροπή. Ένα χαστούκι και στη Μάλτα, στο Κοινοβούλιο. Αυτά συζητούμε συνέχεια. Το, η κυβέρνηση πάντως αρνείται να συγκροτήσει ερευνητική επιτροπή. Και βέβαια στη συζήτηση για το ξύλιμα χρήματος δεν ήρθε ο υπουργό εκείνο. Θα πρέπει να τον καλέσετε εσείς ή να έρθετε στη Μάλτα να του μιλήσετε. Αρνείται επομένως οτιδήποτε, οποιαδήποτε συνεργασία ε, και έχει κλειτευτεί πάρα πολλές φορές από την αστυνομία χωρίς να προκύψει τίποτα. Οπότε βλέπετε ότι αυτή η κυβέρνηση της χώρας μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Λάγκερ. 19... και 20 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε στη Μάλτα με την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, με δικηγόρους, με διαχειριστές ε, περιουσίας, ε, με δημοσιογράφους και ο υπουργό ε, Οικονομικών που προεδρεύει αυτή τη στιγμή στο ΕΚΟΦΗΝ θα είναι εκεί. Λοιπόν, κατόπιν έχουμε την κυρία Μισελ Αντρέα από την Γαλλική Γερουσία. Πού είναι? Ναι, ναι. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για αυτή την συζήτηση. Η καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και στην επίπεδο κινητοποιεί εδώ και πολύ καιρό την αρμόδια επιτροπή της Γαλλικής Γερουσίας και στη συνέχεια αυτού του σκανδάλου για τα Panama Papers αναλάβαμε δράση από τον Μάιο του 2016 για να δούμε τι γίνεται σε μια πάρα πολύ σημαντική γαλλική τράπεζα που έχει μπλεχτεί σε αυτά ε, και ο στόχος είναι να δούμε τι περιθώρια απάντηση υπάρχει, τι γίνεται παρά τα καινούργια ε, μέτρα που υπάρχουν το 2009 γιατί έτσι συγκλονίζεται η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα ε, γιατί μπορεί να έχουμε συνεργασίες ε, και στα πλαίσια του ΩΣΑ αλλά τίποτα στην πράξη δεν αλλάζει. Και τι να βγάλαμε. Είπαμε ότι είδαμε πώς λειτουργεί το σύστημα με κάποιες υπηρεσίες STDR ε, και πρόκειται για κάποια μέτρα τα οποία θέσπισαν οι φορολογικές αρχές της χώρας μας και μετά το 2013 είχαμε πάνω από 47.000 ε, αιτήσει φορολογουμένων και έτσι είχαμε αποζημιώσεις 6,3 δις ευρώ όπου και είδαμε ότι είναι πάρα πολύ ενισχυτικές οι δυσκολίες να δούμε τι γίνεται με τις ε, ρυθμιστικές τραπεζικές αρχές. Δεν υπάρχει συμφωνία ε, μεταξύ των, των διεθνών φορέων για το ποιες είναι οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι υποχρεώσεις αυτών των ρυθμιστικών αρχών στην Ευρώπη. Και συμφωνώ για το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λίστα των φορολογικών παραδείσων. Ακριβώς όπως υποσχέθηκε να κάνει ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και ε, επίσης το, το πώς υπάρχουν εργασίες υπάρχουν και στο website της γερουσίας μας. Υπάρχουν ε, διακρατικές συμφωνίες και το 2011 απορρίψαμε την φορολογική συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Παναμά. Ευχαριστούμε, κύριε Άντρε. Γιώχιμ Πώς από τη Γερμανική Βουλή. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρώπη είμαστε σε ένα κόμβο, σε ένα κεντρικό σημείο καταπολέμησης της ε, φοροαποφυγής, όμως ε, δεν μπορούμε να δράσουμε ε, διότι υπάρχει διχασμός ως προς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Υπάρχουν ε, μοντέλα προστασίας ε, τέτοιων απαντεδόλιων μηχανισμών και η Τερέζα με ο Ντάισελμπλουμ ή ο Γέσοφ Μάσκα, όπως είπε αυτός αυτοαποκαλούμενος σοσιαλιστής δημοκράτης, υποστηρίζουν αυτά τα μοντέλα προστασίας της φοροαποφύγης. Όσο συνεχίζεται αυτό αυτές τις χώρες Μπενελούξ, Μάλτα, Κύπρος. Δεν πρόκειται να μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα και αυξάνεται η δύναμη της ακροδεξιάς και δεν ρυθμίζεται το πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχει προσωπική ευθύνη, ακόμη και από τη δική μου πολιτική οικογένεια δεν επομίζονται τις ευθύνες τους. Συμφωνώ με τον κύριο Κρένερ, δεν υπάρχει κανένας ε, ε, ε, νομικός λόγος που ευσταθεί για την ε, συγκρότηση αυτών των εταιριών γραμματοκιβωτίων. Οπότε ας το απαγορεύσουμε, εν πάση περιπτώσει. Και όχι η Μάλτα, αλλά και το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται από τα υπόλοιπα ε, κράτη-μέλη για φοροαποφυγή. Θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο μαύρος ε, κατάλογος ε, και σε αυτό το μαύρο κατάλογο πρέπει να αναγράφονται και αυτά τα κράτη-μέλη. Μέχρι τότε δεν πρέπει να καταφέρουμε Εγώ Μπορώ να μιλάω εσαΐ, γιατί μιλάμε για ξέπνο βρώμικου χρήματος, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Δεν μπορούμε να δράσουμε και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους νομοταγείς φορολογουμένους, τους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας αυτού και βοηθάμε αυτούς που έχουν αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα με και ξεπλένουν δισεκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπός. Αυτή η πράξη κατά εξουσιοδότηση ε, που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εγκρίναμε εμείς στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα με ειδική πλειοψηφία για ε, συγγνώμη, απορρίψαμε με ειδική πλειοψηφία αυτή την πρόταση ε, για το μαύρο κατάλογο. Ε, τώρα, ευρωβουλευτές, Πίτερ Σίμων από τη Γερμανία. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πόστα από την Ομοσπονδιακή Βουλή. Στην Ευρώπη δεν έχουμε το πρόβλημα μόνο το ότι άλλοι εδώ πέρα κανονίζουν τα φορολογικά μας. Είχε έρθει εδώ πέρα α, ο Υπουργό Οικονομικών της, ε, των Μπαχαμών και μας είπε «Μα τα προβλήματα τα δημιουργείτε μόνοι σας α, ε, οι Ευρωπαίοι, δεν σας θέω εγώ». Και το πρόβλημα είναι ότι έχει δίκιο. Και το δικό μας το πρόβλημα είναι πως υπάρχουν αρκετοί μέσα σε αυτή την αίθουσα που έρχονται από χώρες οι οποίες έχουν ως επιχειρηματικό μοντέλο να κλέβουν τα φορολογικά έσοδα άλλων χωρών. Δεν έχει ούτε μία σχέση με κόμματα και πολιτική τοποθέτηση. Γι' αυτό σας παρακαλώ, τι κάνετε στην Μάλτα. Μιλάμε για κρατικές δομές. Δεν μιλάμε για μικρά πραγματάκια. Όχι. Η Ευρώπη θα διαλυθεί εάν δεν καταφέρουμε να βρούμε κάποια αλληλεγγύη. Και αυτό δεν έχει ε, σχέση με το ότι δεν θέμε φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά όταν, είναι, όταν επιτρέπουν κάποιες χώρες σε πολυεθνικές εταιρείες να πληρώνουν φόρο κάτω από 1% κάτι δεν πάει καλά στην Ευρώπη. Αν λοιπόν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει η Ευρώπη θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις χώρες μας έτσι ώστε να υπάρξει η επικοδομητική συνεργασία εδώ στις Βρυξέλλες. Και το πρώτο βήμα είναι ακριβώς να υπάρχει η αυτόματη πληροφόρηση για τις φορολογικές αποφάσεις που λαμβάνονται. Γιατί αρνούνται μέχρι στιγμή τα κράτη-μέλη να στείλουν τις πληροφορίες στην Κομισιόν των Θεματοφύλακα των Συνθήκων για τις συμφωνίες που υπάρχουν για φοροαποφυγή και γίνεται αγώνας αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες για να φτάνουν όλες οι πληροφορίες στην Κομισιόν. Ε, εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε εμείς να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει εντός της Ευρώπης πριν αρχίσουμε να ασκούμε κριτική εκτός Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε και για το πάθος με το οποίο ε, μιλήσατε. Τα ξέρουμε και στην Επιτροπή. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, ε, θα ήθελα να ρωτήσω τους παρισταμένους εδώ πέρα στο βήμα εάν ε, έχουν κάποιε παρατηρήσει για τις τέσσερις ε, παρεμβάσει που έγιναν ήδη. Καθηγητά, κύριε Πίτ, παρακαλώ. Πολύ σύντομα θα είναι, θεωρώ, πολύ εντυπωσιακό το ότι δεν περιορίζεται στην κατηγόρια, γιατί βέβαια το θέμα είναι παγκοσμίων διαστάσεων. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το τι γίνεται με κάποια σημεία στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιο κοινό παρονομαστή και η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται δεν ομονοεί. Υπάρχουν διχογνωμίε από την άλλη μεριά βέβαια. Υπάρχει και κάποια σύγκληση απόψεων, κάποια σημεία συμφωνία ακριβώ στο θέμα του εντοπισμού αυτών των πραγματικών δικαιούχων, των beneficial owners. Και οπότε είπαμε για το εταιρικό μητρό, πρέπει να γίνουν βήματα προς τα προσοχή με τις ε, απαγορεύσεις. Θέλουμε πρώτα-πρώτα πάντως διαφάνεια. Όλα αυτά παίρνουν νερό, συζητιούνται. Αλλά άπαξ και υπάρξει διαφάνεια, ε, τότε σταματάμε να ε, του στερούμε τέλο πάντων την ελκυστικότητα αυτών των μέρων. Ευχαριστούμε. Ο Νομίζω πως η Ολλανδία πράγματι ιστορικά έχει ένα μέρος της ευθύνης ε, για την φοροαποφυγή, όπως είπε ο Γερουν Ντάισεμπλουμ, η Ολλανδία ήταν μέρος του προβλήματος και τώρα θα πρέπει να γίνει μέρος της λύσης και νομίζω πως ε, η τωρινή μας ε, στάση είναι διαφορετική από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια. Λαμβάνονται μέτρα κατά της φοροαποφυγής σε σχέση με 10 ε, χρόνια πριν. Παραδείγματο χάρη λαμβάνονται πάρα πολλά μέτρα για να γίνει δύσκολη η ζωή, να ανεκνευτούν και να ε, στριμωχτούν οι εταιρείε ε, γραμματοκιβώτια για να σταματήσουν επίσης οι επιθετικές αυτές πρακτικές φόρο αποφυγής και αντιμετωπίζουμε και τους φορολογικούς ε, συμβούλους ε, αλλά πράγματι ε, υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα που πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος ή θέλετε να περιμένετε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, πολύ γρήγορα, λέει ο κύριος Λάκη. Ναι, σε σχέση με αυτό που είπα και εγώ, ότι πρέπει να ταυτοποιήσουμε τα ενίκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτού αρχίσουμε να μιλάμε για την προστασία της φορολογικής επικράτειας κάποιου ε, κράτους μέλους σε σχέση με τις εξωτερικές ε, απειλές ε, των, των ε, διεθνών οικονομικών ροών, να τις προστατεύσουμε από τη δράση των φορολογικών παραδείσων. Ε, ναι, μιλήσατε για τις ε, πρακτικές των κρατών. Ναι, πρόκειται για επιθετικό φορολογικό ανταγωνισμό ε, που αφαιρούν φορολογικά εισοδήματα από κάποια κράτη-μέλη και όντως μπέψα η φορολογική εναρμόνιση. Αυτός ο δρόμος πρέπει να ακολουθήσουμε και φορολόγηση των πολυεθνικών. Αλλιώ ε, θα ε, είναι άκρατο αυτό ο φορολογικό ανταγωνισμός και θα καταστραφούν τα δημόσια οικονομικά. Η φορολογική βελτιστοποίηση, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμό είναι αυτά που χρειαζόμαστε, ούτω ώστε να, αποκτή, να ανακτήσουν την κυριαρχία του οι δημόσιε οικονομικέ αρχέ. Θέλετε κι εσεί να μα πείτε κάτι. Ναι, ναι, δύο προτάσει. Καλή μαύρη κατάλογη. Και η γκρίζη μας, ε, μας βοηθάει γιατί έχουμε και το τραπεζικό απόρριτο και θα γίνουμε πιο πολιτισμένοι. Ε, και έτσι μπορούν να αποφευχθούν οι μεταφορές ε, αυτών των υπέρογων ποσών. Συνήθω δεν συμφωνώ με τον κύριο Πόσα από το Γερμανικό Κοινοβούλιο, σήμερα που πρέπει να το ομολογήσω. Ευχαριστούμε. Ο Μίγουελ Τιάγκο από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Πού είστε κυρία μου? Eh, Ευχαριστώ. Θέλω... Από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας είμαι. Ε, ε, είμαι βουλευτής ε, στη στο, στο Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας και μετέχω στην Εξεταστική Επιτροπή. Σε τρεις εξεταστικές επιτροπές για αυτά τα ζητήματα. Ε, υπάρχει κοινό ε, παρονομαστής ε, αποκεφαλοποίηση των τραπεζών, επτώχευση των τραπεζών. Σχετίζεται αυτό βεβαίως με τη συζήτηση τη σημερινή για τις υπεράκτιες εταιρείε, φορολογικούς παραδείσους, ε, δηλαδή χώρες με ε, πιο ευνοϊκά ε, φορολογικά συστήματα που χρησιμοποιούν μεγάλες επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο για την φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη, το ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματος και ξέρουμε ότι πλήττονται τα συμφέροντα των υπόλοιπων κρατών μελών. Μία πρώτη παρατήρηση. Ε, φαίνεται σαν ξένο σώμα η offshore εταιρεία σε σχέση με το κεφάλαιο, μα είναι μέρος του μεγάλου κεφαλαίου. Γιατί το παρουσιάζουμε έτσι. Και ε, λαδώνει το, το, το, μηχανισμό ε, του, του, κεφαλαίου. Ας, αφήσουμε αυτές τις ηθικολογικές συζητήσεις. Δεν είναι ξένο σώμα η offshore εταιρεία. Ε, οι μεταφορές προς τις offshore, ο εντοπισμός ε, των πραγματικών δικαιούχων, ο έλεγχος ε, των λογαριασμών. Μα τι λέμε τώρα, θέλουμε να αφήσουμε το λύκο να φλέει τα πρόβατα, αστειευόμαστε σίγουρα. Ε, δεν δηλώνουν όπως θα έπρεπε ούτως ή άλλως οι τράπεζες στις μεταφορές προς τους λογαριασμούς των offshore. Ε, τα εθνικά συστήματα, ναι, το κάθε κράτος έχει το δικό του σύστημα. Έχουν προταθεί ε, διάφορες λύσεις. Δεν υπάρχει όμως πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις. Τα είπαμε ήδη να φορολογούνται οι εταιρείε, όχι σε σχέση με τα φορολογικά εισοδήματα, αλλά σε σχέση με το κομμάτι του τζίρου που το, ε, τοποθετείται, που καταλογίζεται σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ε, η καταγραφή των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών με τις υπεράκτιες, ε, η ε, εξωτερικοποίηση, το τη καταγραφή των φορολογικών εσόδων από διαφορετικές ε, δικαιογορικές ε, εταιρείε. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση. Διακόπτει ο Πρόεδρος τώρα από την Ελλάδα. Κύριος Αθανασίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είχα ετοιμαστεί να πω δύο λόγια για τα Panama Papers δεν θα μπορούσα να πω τίποτα καλύτερα από αυτό που ανέφερε το μέλος της Bundestag Herr Αλλά ο καθηγητής Πιτ είπε δύο λέξεις που με έπεισαν ότι κάνουμε ένα αθέλητο λάθος. Ποιο είναι το λάθος. Χρησιμοποιούμε μια αλήθεια για να κρύψουμε μια άλλη αλήθεια. Και ποιες είναι οι δύο λέξεις του καθηγητή Πιτ που με έπεισαν γι' αυτό. Οι λέξεις βρώμικο χρήμα. Dirty money. Εάν το θέμα μας σήμερα δεν ήταν τα Panama Papers, αλλά το βρώμικο χρήμα, δείτε τι θα μπορούσε να συμβεί. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής η Apple και η Amazon, αμερικανικές εταιρείες. Ναι, που σχετίζονται με τα Panama Papers. Το έχω διερευνήσει, ήμουν 40 χρόνια δημοσιογράφος το έχω διερευνήσει και προσωπικά. Αν όμως ο τίτλος της σημερινής συζήτησης ήταν «Dirty Money», βρώμικο χρήμα, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για την Deutsche Bank, παραδείγματο χάρη. Γίνεται μια δίκη αυτέ τι ημέρε στο Μιλάνο. Οι Ιταλοί συνάδελφοι θα μπορούν να μα πούν ε, κάτι. Το business Bloomberg την περασμένη εβδομάδα κάτι έγραψε. Και τι έγραψε. Δεν μπορώ να συζητώ για τα Panama Papers και να μην συζητώ αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα ε, στο Μιλάνο και δημοσιεύεται στο business, Bloomberg Business Week 10 δισεκατομμύρια δολάρια η τράπεζα αυτή δεν τα ενέγραψε στα βιβλία της. Όταν μια μεγάλη τράπεζα, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που δίνει το στίγμα της Ευρώπης, δεν γράφει στα βιβλία της 10 δισεκατομμύρια δολάρια και δημοσιεύεται στο business Bloomberg, εγώ δεν μπορώ να σιωπήσω. Αν το θέμα μας ήταν dirty money, καθηγητά Πιτ, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμη ακόμη και για τη Volkswagen, ένα μέλος της οποίας έχει συλληφθεί στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και αλήθεια, δεν είμαι εκτός θέματος αν πω Είμαστε κατώτεροι οικολογικά στην Ευρώπη από τις Ηνωμένε Πολιτείες Δηλαδή οι εκπομπές ρήπων στην Ευρώπη πρέπει να είναι να μην τιμωρούνται ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείες να τιμωρούνται. Η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο το ανέχεται αυτό. Θα μπορούσαμε... Time is over. Please. Είναι ενοχλητικό, τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα. Ε, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνογερμανικής Φιλίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αγαπώ την ε, Γερμανία και δεν τα λέω από κακία από αυτό. Δεν, δεν έχω καμία πρόθεση. Αλλά, και τελειώνω με αυτό, ε, κύριε Πίτ, συναντηθήκατε με, με τον Τζόζεφ Στίγκλιτς και συζητήσατε για τη σκιώδη οικονομία, τη shadow economy. Ελπίζω να συζητήσατε μαζί του και για τα δημόσια χρέη των χωρών της Ευρώπης. Πληθυντικό χρησιμοποίησα. Διότι χθε μνημόνευσα τον Τζόζεφ Στίγκλιτς και τον Πολ Κρούγκμαν και ο κύριος Ντομπρόφσκης απέρριψε ε, τις θέσεις των οποίων αντέγραψα και το ανέφερα. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη so, που υπερεύει okay. το χρόνο. Dank. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά είχαμε πει, εντάξει. Ε, ξεπεράσατε λίγο το χρόνο. Λοιπόν, 9 Φεβρουαρίου στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητήσουμε και τα των τραπεζών και μεμονωμένων τραπεζών. Οπότε θα, θα ακουστούν και αυτά. Δεν έχουμε πιάσει ακόμα την ε, Deutsche Bank, αλλά θα έρθει ο σύνδεσμος των γερμανικών τραπεζών, θα εκπροσωπηθεί εκεί πέρα. Με τον πρόεδρό τους νομίζω. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Μαρτ Φαντεβέν από την Ολλανδική Γερουσία. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τι μας είπαν οι εμπειρογνώμονες και μπράβο. Μπράβο στα όσα είπανε παρόλα αυτά. Όμω, παραλείψαμε μία εξέλιξη Στι 11 Δεκάτου του 2016 το Συμβούλιο της Ευρώπη δέχτηκε το ψήφισμα 21-30 που αφορά τα Panama Papers και από πλευρά τη Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων είχαμε μια γνωμοδότηση πάνω σε αυτό το ψήφισμα και είχα γνωμοδοτήσει και εγώ σε σχέση με αυτή την γνωμοδότηση και λέμε ότι θα πρέπει το Συμβουλίο της Ευρώπης με τον ΩΣΑ να συντάξουν κάποιους κανόνες όσον αφορά την έμεση φορολογία και όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού αυτών των εταιριών offshore και έτσι να μπορούμε να ε, παρακάμψουμε αυτούς οι οποίοι στείνουν ε, τα κόλπα αυτά. Θα ήθελα να μου πούν οι εμπειρογνώμονες τι πρεσβεύουν όσον αφορά αυτή την ε, πρόταση για να μπορέσουμε να ε, απαλλαγούμε από αυτήν την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Ευχαριστώ. Κατόπιν ο Λουί Μισελ από το Βέλγιο Ευρωβουλευτής. Oui, Μάλιστα, Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα τις ευχαριστίες μου προς ε, όλους τους προσκεκλημένους. Εγώ θέλω τώρα να συζητήσουμε το εξή συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίω και συμφωνώ με αυτή την ε, αγανάκτηση σε σχέση με αυτό το αφόρητο φαινόμενο και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να κάνουμε αυτή τον, ε, την αγανάκτηση, να την κάνουμε πολιτική βούληση και αυτό να ισχύσει για όλα τα κράτη. Ε, φυσικά είναι πολιτικό το θέμα στην τελευταία ανάλυση. Και έχω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς τι πληροφορίες μπορέσατε να έχετε όσον αφορά τα κριτήρια της due diligence για τους ενδιάμεσους της δέουσα επιμελίας. Τι γίνεται με τις εθνικές αρχές που ελέγχουν ε, και θα πρέπει αυτός ο έλεγχος να γίνεται σε ε, όλη την διαδρομή που ακολουθούν αυτοί που διαπράττουν αυτή την απάντη. Και τι δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια αντίστοιχη υπηρεσία πανευρωπαϊκή, ούτως ώστε να ελέγχει καλύτερα τις ύποπτες ροές, ε, γιατί αυτό γίνεται παντού στην Ευρώπη και είναι διασυνοριακό. Για πέστε μας επίσης, έχουμε την ΦΑΤΚΑ στην ε, ε, Αμερική. Δηλαδή έχουμε την υποχρέωση των Αμερικανών που θα πρέπει να δηλώνουν στις ε, αρχές το σύνολο της περιουσίας που έχουν και στο εξωτερικό. Οπότε μήπως θα μπορούσαμε και εδώ να έχουμε ένα τέτοιο φορέα ή ένα τέτοιο θεσμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Πιτ, στην απάντησή σας επίσης αναφέρατε, γιατί και άλλοι το ανέφεραν, το ότι συχνά προσφεύγει ο κόσμος σε ελβετούς δικηγόρους. Μήπως θα μπορούσατε να μας τα πείτε πιο συγκεκριμένα ακριβώς για ποιους λόγους υπάρχει ακριβώς αυτή η ζήτηση για τους ε, ε, ελβετούς δικηγόρους. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Ε, επίσης, θα ήθελα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, τι ορισμός μπορεί να υπάρξει ο ορισμός φορολογικής απάτης και φοροαποφυγής. Συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι πολλές φορές η διάκριση είναι δύσκολη ή ανύπαρκτη. Ότι δηλαδή η... πολλές φορές βαφτίζεται το παράνομο νόμιμο. Πάνω σε αυτό αν γίνεται να εμβαθύνουμε. Äh, äh, κύριε Μισελ, για τις δύο τελευταίες συγκεκριμένες ερωτήσεις, ε, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Πίτ. Um, Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτα απ' όλα νομίζω πως μία ερώτηση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Αφορά το ερώτημα το 13 που μου είχατε θέσει για τους Ελβετούς δικηγόρους στην Γενέβη. Πώς τυχαίνει να υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση ε, δικηγόρων που είναι, θα έλεγε κανείς, ε, ο βασικός διάβλος για τα Panama Papers. Μα τα Panama Papers είναι ένα τυχαίο παράδειγμα, μια ματιά στην σκιώδη οικονομία. Υπάρχουν πολύ περισσότερα γύρω από αυτό και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούσαν. Και ακριβώ αυτό εννοούσα όταν μιλούσα για την παραδοσιακή νομική δουλειά και το ότι γίνονται οι δικηγόροι οικονομικοί παράγοντες και υπάρχει μια ευαίσθητη γκρίζα ζώνη δηλαδή αν κάποιος παραδείγματο χάρη εκτελεί μια διαθήκη μπορεί πράγματι για λίγο καιρό να είναι διαχειριστής αυτό είναι το παραδοσιακό. Αλλά αν αρχίσει να δημιουργεί δομές, ε, υπεράκτιες εταιρείε ε, κτλ. και να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, ε, αυτό ανήκει θα έλεγα στον τομέα του οικονομικού δρόντος. Στην τωρινή βεβαίως ελβετική ερμηνεία δεν εμπίπτει εκεί. μάλιστα περίφθη το αίτημα αλλαγής του νόμου από το Ελβετικό Κοινοβούλιο και αυτό ακριβώς αφορά το ερώτημα 13 που μου έχετε θέσει εδώ. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να κάνω είναι να σας ε, ενθαρρύνω να κοιτάξετε την κατάσταση στις δικές σας ε, χώρες, αν διαφέρει, και το διαχωρισμό που κάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αν μου επιτρέπετε δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με τον Έλληνα συνάδελφο ότι είναι ευρύτατο το θέμα και αφορά και τους φόρους και το ξέπλυμα χρήματος και ίσως και άλλα ζητήματα. Ένα άλλο θέμα, οι μαύρες λίστες αναφέρθηκαν και πράγματι τώρα βρίσκεστε σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί συνειδητοποιείτε και οι ίδιοι ότι είστε μέλος, μέρος, είμαστε θα έλεγα μέρος του προβλήματος. Οι μαύρες λίστες είναι δύσκολες αν είναι κάποιος ο ίδιος μέρος του προβλήματος, οπότε πρόταση η πείρα μου από τα 25 χρόνια στον ΩΣΑ που ήμουν αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμφωνήσαμε, συμφωνούσαμε σε έναν κοινό παρονομαστή. Και μετά το ερώτημα είναι εάν το στέλναμε στις χώρες και λέγαμε πρέπει να το εφαρμόσετε ή εάν υπήρχε μια υπερεθνική μονάδα οικονομικών πληροφοριών. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Αλλά αυτό το οποίο κάνουν είναι κάτι το οποίο ξέρετε κι εσείς εδώ πέρα παρακολουθούσαν την συμμόρφωση των χωρών σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα. Και μετά, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο συμφωνούν όλοι, τότε μπορούμε να πούμε ότι ναι, κοιτάμε την εφαρμογή και υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες ε, δεν συμμορφώνονται. Αυτό έκανε το FTA, Financial Action Task Force, και τότε γράφεις μια μαύρη λίστα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ποιο είναι πρώτος, Γκρότε και Λεωγιέ. Ναι, δύο σημεία σύντομα. Πρώτα απ' όλα για την ε, άμεση φορολόγηση σε κονδύλια που πηγαίνουν ε, σε φορολογικούς παραδείσους. Ε, εμείς στην Ολλανδία είπαμε ότι θα ήταν καλή μια ευρωπαϊκή κίνηση για να γίνει κάτι τέτοιο ε, μέχρι στιγμής ε, δεν έχει υπάρξει κάποια στήριξη για να κάνει κάτι τέτοιο μόνη της η Ολλανδία. Δεύτερον, για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ολλανδία κάτι ανάλογο με την ΦΑΤΚΑ. Κοιτάξτε, η ε, νομίζω ότι υποτιμούμε τις ε, δυνάμεις μας. Εάν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί, πρέπει να έχουμε και εμείς την δυνατότητα, νομίζω, να το κάνουμε. Μπορεί να γίνει μέσω των εκθέσεων ανά χώρα, να ε, επιβάλλουμε κυρώσει στι πολυεθνικές οι οποίες δεν συμμορφώνονται. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να υποτιμούμε αυτούς τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λαουρέ. Ναι, για να απαντήσω και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις ε, του ε, αξιότιμου κ. Μισελ. Η Ben Paribas Reportis, η NG, KBC, Dexia, οι μεγαλύτερες δηλαδή τράπεζες του Βελγίου και κάποιες άλλες διαχείρισεις χαρτοφυλακίου μας είπαν ότι ουδέμια σχέση έχουν με τη διεθνή φορολογική απάτη. Ότι όλα καλά έχουν εξηγιάνει τα οικονομικά τους, γιατί είχαν περισσότερες θηγατρικές ε, στα φορολογικούς παραδείσους. Τους ρωτήσαμε με, ε, για τις εσωτερικές διαδικασίες που χρησιμοποιούμε και έφτιαξα εγώ ένα data room, ε, επειδή τώρα έχουν όλες οι ειδικές διαδικασίες Φτιάξαμε αυτό το data room και όλοι μπορούν να βλέπουν τις ιστορικές διαδικασίες που ακολουθούν αυτές τις τράπεζες. Το συμπέρασμα είναι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να τις προφυλάξουμε από τον πειρασμό να, για να μην υποτροπιάσουν στο μέλλον. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε ε, ε, διεθνείς εφορολογικούς δόλιους μηχανισμούς εάν πρώτον δεν έχουμε τη φαιά ουσία που φτιάχνει αυτό το μηχανισμό και δεύτερον αν δεν έχουμε ένα οικονομικό κύκλωμα και γι' αυτό οι νομοθέτες για τα οικονομικά θα πρέπει να εστιάσουν προσοχή τους αυτά τα δύο σημεία. Λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι παρότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει να γίνουν περισσότερα για τον εντοπισμό αυτών των μηχανισμών για τη διεθνή απατή. Δεν εφαρμόζεται αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει επίγνωση όμως και έχουν κατατεθεί προτάσεις για την αναβάθμιση του νομικού πλαισίου. Δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, μόνο να πω ότι φυσικά συμφωνώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μια υπεραρχή ε, για την ιδίωξη οικονομικού εγκλήματος για την δίωξη της φορολογικής απάτης κυρίως φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστούμε. Κύριε Κράνερ, ε, όχι υποχρεωτικά, αλλά άμα θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Ε, λέτε ότι δεν πρέπει να υποτιμά τη δύναμή της η Ευρώπη και θα πρέπει να κάνει περισσότερο. Μα το κάνουμε, συνεργαζόμαστε. Ε, εάν δεν προσπαθεί ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου όμως. Αυτή είναι η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όχι ανταγωνισμός ε, διακρατικός. Αυτό ε, θα μας δώσει περισσότερη δύναμη και έτσι θα αποφύγουμε αυτό τον ποδέστρο ρόλο που έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε για αυτή την έκκληση που απευθύνατε σε όλους. Άλλους τρεις ομιλητές, Αρνόλτ Μέρκης από την Ολλανδία, από τη Γερουσία, από το νοσόμα. Από το κάτω σώμα, συγγνώμη. Ναι, πολύ ωραίο το, το προφέρετε αυτό το τβέιντε camera. With, uh, at um... Της Βουλής δηλαδή, όπου εργάζομαι. Μας έχουν επικρίνει και δικαίως. Ξέρετε και στο δικό μας κοινοβούλιο επικρίνουμε εαυτούς αυτούς ακριβώς διότι το, η κυβέρνηση της χώρας προσπαθεί να αναβάλει την υλοποίηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, την ε, άσκηση της φοροδιαφυγής και προσπαθεί η κυβέρνηση μέχρι το 2024 να αναβάλει την εκτέλεση αυτής της πρότασης. Εμείς όμως ως Κοινοβούλιο είπαμε δεν θέλουμε την αναβολή και απορρίψαμε την κυβερνητική πρόταση. Άρα θέλω να γνωρίζω ότι όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να βολεί, εμεί όχι ω κοινοβούλιο. Έτσι πρέπει ο ένα να διδάσκει τον άλλον τι πρέπει να γίνει. Άρα θα πρέπει κανείς να θέτει τα σωστά ερωτήματα προς την κυβέρνησή του. Τέλος πάντων, ταυτόχρονα συζητούμε και για τη φοροαποφυγή και για την φοροδιαφυγή. Τα συζητάμε μαζί αυτά και κάπως τα μπερδεύουμε. Τέλος πάντων θέλω να σας πω για την list, για τη μαύρη λίστα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστός ορισμός. TST, μαύρη λίστα. Αν δεν πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποια χώρα που έχει πολύ λίγους, πολύ χαμηλούς ε, φόρους, δεν είναι φορολόγιος παράδεισος, ε, τότε έχουμε πρόβλημα. Άρα τουλάχιστον ας υπάρχει ένα ελάχιστο ένα μήνυμα, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Φορολογικούς παραδείσους, προτιμησιακά καθεστώτα κλπ. Άρα, ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον ορισμό, αλλιώς θα γίνει κάτι σαν το, αυτό που έγινε στο παρελθόν με τον ΟΣΑΒ, που είχε τη μαύρη λίστα. Αλλά δεν έβρισκε καμιά χώρα και κανένα φορολογικό παράδεισο σε αυτή τη μαύρη λίστα. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Άλλου 9 έχουμε στον κατάλογο και 25 λεπτά. Και θέλουμε να κάνουμε και ένα τελικό γύρο, να ακούσουμε δηλαδή τους ε, υπηρογνώμονες. Η Νέσης Μόνκης ε, από την ε, Λετωνία. Πού είστε? Γεια, Λαμπρίτ, κολέγγι. Βέλος, Ευχαριστώ. Εμείς υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φοροαποφυγή και την καταπολέμηση του, της νομοποίησης παρανόμων εσόδων. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 700-800 υπεράκτιες. Είναι μικρή όμως οι οικονομία, είναι τεράστιος αυτός ο αριθμός. Ε, πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη ρύθμιση για την ε, ε, κατανομή των φορολογικών εσόδων και μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρηματίες φτιάχνουν την προσθεμένη αξία. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν της, των δικών μας εργασιών και της κυβέρνησης. Μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων και βελτίωση του επιχειρηματικού κλίμα, κλίματος. Βλέπουμε όμως, διαπιστώνουμε και πάλι ότι Υπάρχουν αντικρούμενα συμφέροντα. Ε, ελπίζουμε ότι οι κανόνες του ΩΣΑ θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε το ξέπνο βρώμικου χρήματος. Ε, ξέρετε ότι, ε, όπως είπαν και πολλοί ομιλητές, ε, η νομοθεσία προβλέπει πως φορολογείται η εταιρεία για το κομμάτι του τζίρου στη χώρα όπου έχει καταλογιστεί λογιστικά. Ε, λοιπόν, ε, θέλω να ρωτήσω, σε ποιο σημείο τώρα έχουμε φτάσει για την ε, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τα φορολογικά στοιχεία και τις φορολογικές ε, συμφωνίες, αυτά τα tax rulings. Θα πρέπει ανάμεσα στα κράτη-μέλη να υπάρχει συστηματική ανταλλαγή. Εάν όχι, Εσπευσμένα θα πρέπει να εφαρμοστεί η ρύθμιση αυτή. Είναι κέρια σημασίας. Μπορούμε να μιλάμε μόνο γι' αυτό χωρίς πλήρη εφαρμογή, αλλιώς δεν πρόκειται να έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Τώρα... Ο κύριος Μπονίτσι από τη Μάλτα είναι ο τελευταίος ομιλητής από Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Έχω διατελέσει υπουργό και τώρα ως υπουργό προεδρεύω και του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη και του Συμβουλίου Υπουργών ε, Πολιτισμού. Είμαι βέβαια μέλος του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας πω τα εξή Σε τρεις άξονες θέλω να σας εξηγήσω σε σχέση με όσα ακούσαμε ότι πρώτα πρώτα έχουμε το έργο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ε, και ναι ναι ναι ε, κοντός κοντός είμαι σύντομο, <laughs> κατά κάποιο τρόπο σύντομα θα σα τα πω οπότε πρώτα πρώτα τι έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, όσον αφορά αυτές τις ε, αποκαλύψεις από τον Παναμά και να δούμε τι θα μας πούνε οι ειδικοί για αυτή την ε, τριπλή προσέγγιση. Πρώτα πρώτα έχουμε την οδηγία για το ξέπλυμα και ελπίζω η Προεδρία μας να ολοκληρώσει αυτή τη διαδρομή, να κλείσει με, πολιτική συμφωνία πριν το καλοκαίρι. Δεύτερον έχουμε την οδηγία όσον αφορά την αντιμετώπιση ε, μέσω του ποινικού δικαίου και ε, το έχουν συζητήσει οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, υπάρχει ευρεία συνένεση και στην ε, Μάλτα κάναμε το άτυπο συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και επίσης υπάρχει ο κανονισμός της αμοιβίας αναγνώρισης όσον αφορά κατασχέσεις κλπ. Και αυτό επίσης το ήταν με θετικό μάτι οι Υπουργοί την περασμένη εβδομάδα στην πατρίδα μου. Τώρα κάτι άλλο για κάποιες παρατηρήσεις που άκουσα από τον συνάδελφο της αντιπολίτευσης. Ε, πάντα τίνει στην μικροπολιτική, τέλος πάντων και την κομματική ε, ε, αντιμετώπιση, αλλά νομίζω ότι θα τα πούμε καλύτερα στην Βουλή μας. Τώρα το τρίτο θέμα που θέλω να σας πω είναι άκουσα για την Μάλτα για ε, τα χρηματοοικονομικά μας από κάποιους ε, ευρωβουλευτές. Σας διαβεβαιώ ότι το σύστημά μας είναι αποτελεσματικό, υγιές και στεγανό. Δεν συμφωνώ ότι είμαστε κάποιο είδου παράδεισος offshore. Διαδοχικές κυβερνήσεις στην χώρα επί πολλά χρόνια το εξασφάλισαν ότι εμείς έχουμε σύστημα το οποίο ε, συνάδει με την ε, νομοθεσία. Αποκρούει μάλιστα τα επιχειρήματα περί του αντιθέτου. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται εκλογικό αγώνα. Ε, στη, στη Μάλτα μπορείτε να το κάνετε. Από τους ευρωβουλευτές έχω τους ομιλητές ε, και σας λέω, έχουμε 20 λεπτά και θέλουμε το τελευταίο να μιλήσουν οι εμπειρογνώμονες. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να μην υπερβείτε το χρόνο αγόρευσης. Ντάριος Ροζάτη, Φάμπιο Ντεμάση, μετά Γιάννη Κόφε, ένας από τους συνεισηγητές ε, και ούτω κάθε εξής. Ντάριος, συντονιστής του ΕΛΚ στην Επιτροπή Πάνα. Ευχαριστώ τους, τα μέλη του πάνελ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψει τους, γιατί είναι φλέγον το ζήτημα της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Δύο ερώτησεις έχω. Πρώτα προς τον κύριο Πιτ. Αλλά και οι υπόλοιποι μπορούν να απαντήσουν, βεβαίω. Όλοι τόνισαν πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο των διαμεσολαβητών, αυτών των intermediaries για την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Ποιοι είναι αυτοί οι διαμεσολαβητέ, ε, δικηγορικά γραφεία, φορολογικοί σύμβουλοι, λογιστές, αλλά και τράπεζες φυσικά. Οι τράπεζες ε, υπάρχονται σε ρυθμίσεις. Όλες οι υπόλοιπε ομάδες όμως υπάγονται σε αυτορύθμιση, κάτι κώδικες διοντολογίας έχουν και τέτοια. Λοιπόν, ε, αρκεί αυτή η αυτορύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για αυτούς τους διαμεσολαβητές για να σταματήσουν να διευκολύνουν και να επικουρούν ε, για τη διοχέτευση αυτών των ε, παρανόμων ε, ροών εσόδων προς υπεράκτους λογαριασμούς. Πώς χρειάζεται εξωτερική ρύθμιση του κράτους για αυτά τα επαγγέλματα, τουλάχιστον για κάποιες από αυτών των επαγγελμάτων. Δεύτερον, σε σχέση με τις ΙΠΑ, αυτά που ξέρουμε για τις ΙΠΑ, γιατί ακούσαμε και σε διάκροασεις της ΠΑΝΑ ότι ε, κατάφεραν να περιορίσουν το μέγεθος της φοροαποφυγής φοροδιαφυγής με την εισαγωγή του περίφημου, της περίφημης νομοθεσίας FATCA. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό ισοδύναμο της νομοθεσίας ΦΑΤΚΑ. Μήπως θα ήταν ένα καλό βήμα για την καταπλώση αυτών των πρακτικών. Ευχαριστούμε κύριε Ροζάτη. Ε, Φάμπιο Ντεμάζη, αντιπρόεδρος ε, της ΠΑΝΑ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τη Μάλτα δεν έχω πολλά σχόλια. Κατά κανόνα όταν κάποιος εκπρόσωπος ε, κυβέρνησης λέει η χώρα μου δεν είναι φορολογικός παράδεισος συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Τέλος πάντων. Ε, συμφωνώ με πολλές από τις εκτιμήσεις των συναδέλφων και ε, πράγματι σωστά αυτά τα οποία ακούστηκαν. Έχουμε τα φορολογικά καρτέλ ε, στην Ευρώπη, έχουμε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και το offshore από ό,τι φαίνεται είναι το modus operandi, έτσι λειτουργεί ε, η οικονομία σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος από την Αυστρία, αλλά η αυστριακή κυβέρνηση και η γερμανική κυβέρνηση είναι κατά της ε, δημοσιοποίησης τέτοιων στοιχείων γιατί λένε ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα. Δύο ερωτήσεις τώρα στον κύριο Πίτε. Έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό τον ε, καιρό μια συζήτηση για το ότι τα καταπιστεύματα για την κληρονομιά θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημοσιότητας γιατί αφορούν μόνο κληρονομίες Ποια είναι η θέση σας για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είναι ε, γνωστά τα ονόματα των ιδιοκτών και κατόπιν ε, με την εμπειρία που είχατε από το Financial Action Task του ΩΣΑ. Είχαμε εδώ πέρα, απορρίψαμε μάλλον πρόσφατα την μαύρη λίστα των ε, χωρών για ξέπλυμα χρήματος γιατί δεν περιείχε τον Παναμά, τις και τις υπόλοιπες χώρες και τι τι γίνεται τελικά. Από ό,τι φαίνεται εμείς ε, το απορρίψαμε, αλλά και να το είχαμε περάσει δεν γίνεται τίποτα. Το ε, παίρνουν, το διαβάζουν και μετά πάνε στη δουλειά τους, πάνε για καφέ κτλ. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα έπρεπε να κάνουμε τις δικές μας αναλύσεις εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν χρειαζόμαστε και κάποια εργαλεία, κάποιες κυρώσεις για ε, αυτούς οι οποίοι λειτουργούν από αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστώ η συνεισηγητριά μας, ε, ο συνεισηγητή μας τώρα, με συγχωρείτε, ο κύριο Κόφοντ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο πρώτα απ' όλα. Ε, θα πρέπει... Όταν μιλάμε για να ξαναδώσουμε αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη ίσως είναι μια καλή ιδέα γιατί βλέπουμε ότι η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέε ευκαιρίε και για του θερμοκράτε και για όσους προσπαθούν να αποφύγουν τη φορολογία κτλ. Παραδείγματο χάρη σήμερα είδαμε ένα πρόστιμο ρεκόρ, μισό δισεκατομμύριο δολάρια, το οποίο επιβλήθηκε. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν συνεχώ και πρέπει να ενισχύσουμε και την νομοθεσία και στι χώρε μα, Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο είπε ο Λουί Μισελ, δηλαδή να έχουμε μια ευρωπαϊκή μονάδα ε, οικονομικών πληροφοριών, γιατί έχουμε συζητήσει εδώ πέρα με τις διοκτικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ε, κρατών μελών, μεταξύ των διοκτικών αρχών. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, μιλάμε για την φοροαποφυγή Έχουμε την κώδικα συμπεριφορά στη σχετική ομάδα ε, για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, αλλά δεν λειτουργεί γιατί τα κράτη-μέλη εργάζονται με μυστικότητα, με ομοφωνία και δεν μπορούν να απαγορεύσουν ακριβώς ε, τέτοια ε, διασυνοριακές πρακτικές. Γι' αυτό ακριβώς συζητήσαμε τα panet boxes. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ε, αναγκάσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην ε, ομάδα για τον κώδικα συμπεριφοράς να κάνουν κάτι. Και τέλος, συμφωνώ με τον αυστριακό συνάδελφο, η διαφάνεια, η αποτελεσματική συνεργασία, η δίκαιη φορολογία, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ε, μπουν στο προσκήνιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τον Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους ε, για τις παρεμβάσεις τους. Ε, τα ταπορίσματα των εξεταστικών επιτροπών ε, και οι συστάσεις σας θα μας βοηθήσουν για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στο Συμβούλιο. Ερωτήσεις. Μετά από όλες τις αποκαλύψεις μπορείτε να μου πείτε πόσους φακέλους ερευνούν οι φορολογικές αρχές. Και επειδή μιλήσαμε για διάφορα οικονομικά συμφέροντα για τις ε, τράπεζες και τις Big Four, που είναι ε, και δικαστές ε, και κατηγορούμενοι, γιατί μιλάμε για τις κυβερνήσεις, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τους κατόχους υπερακτίων λογαριασμών, δεν πιστεύετε από όσα έχετε ακούσει ότι θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων. Και τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιο είναι το πλέον επίγον που πρέπει να γίνει για να συνεργαστούμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο Μίγουελ Βιέγκας, ο ευρωβουλευτής μας από την Πορτογαλία. Πού είστε? 142 ε, εκεί είσαστε μάλιστα. Θα ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για τα ε, εθνικά ε, συμφέροντα που τελικά περιορίζουν ε, το ποσοστό των φρολικών εσόδων που θεωρείται ως καταγραφή στο Βέλγιο. Είναι πολύ γνωστή η πρακτική το πλαίσιο της καταπολέμησης φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, ε, τι πιστεύετε μπορούμε να φανταστούμε να ε, καταργηθεί αυτό το προνόμιο του Βελγίου και να αποφύγουμε την εκτεταμένη χρήση αυτή της πρακτικής και σε άλλες φορολογικές επικράτειες. Μια, δύο ερωτήσεις προς του, τα μέλη του πάνελ. Ε, ως προς τη μεταφορά των ε, οδηγιών σε εθνική νομοθεσία, ξέρετε υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, ε, όταν μιλάμε για μετρητά, μόνο πάνω από 5.000 ελβετικά φράγκα υποχρεούστε να κοινοποιήσετε τα στοιχεία και γι' αυτό μιλάω για τη μεταφορά των οδηγιών στην εθνική νομοθεσία. Τι πώ μπορούμε να φύγουμε από αυτό το περιθώριο ελιγμών. Επίσης μιλάμε για τους πραγματικούς ε, δικαιούχους. Από ποιο επίπεδο και μετά θα πρέπει να τους ε, εντοπίζουμε και κατονομάζουμε 25%. Εγώ ξέρω ότι ακόμα και 5% θα μπορούσαμε να αποφύγουμε για να ελέγξουμε μια επιχείρηση. Λοιπόν, μήπως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το κατόφλι και άρα να καταστήσουμε και το μέτρο αποτελεσματικότερο. Ευχαριστούμε. Άλλοι τρεις ομιλητές. Παρακαλώ σύντομοι να είστε όλοι. Ε, Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη εκδήλωση κατά την οποία ανταλλάσσουμε απόψεις. Αλλά δεν αρκεί μία φορά να γίνεται αυτό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε περαιτέρω, διότι το θέμα της καταπολέμησης φοροδιαφύγης και φοροαποφυγής είναι ε, κάτι το οποίο καταγνεί το πόσο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να εμβάσει ένα σωρό λεφτά από τη μια γωνιά του κόσμου στην άλλη. Άρα θα πρέπει και κάποιο να ανέβει επίπεδο για να δώσει σωστέ απαντήσει. Και συμφωνώ με τον ε, κύριο Κράινερ. Πώ να τον ανεβιώσιμη η Ένωση όταν ε, ε, βρισκόμαστε σε κάποιον ανταγωνισμό της εξίσωσης προς τα κάτω, τέλος πάντων το, το, το ποιος θα φοροδιαφύγει περισσότερο. Προσοχή, γιατί κάποιε εταιρείε πλέον 0,005 του όσο θα έπρεπε. Ε, αυτό είναι απόδειξη του ότι έχει αποτύχει το σύστημα. Πώ είναι τον να δεχτούμε η κυβέρνηση ε, πάρα πολύ κοντά ε, σε εδώ στο κοινοβούλιο ε, να, να, να και άλλα να εξαγγέλει και άλλα να κάνει. Γιατί πρόκειται για χρήματα που είναι πολύτιμα για του πολίτε μα. Ναι, ναι, ναι, τώρα τελειώνω, Πρόεδρε, και αυτό σα ε, τονίζω ότι η ευρωπαϊκή διάσταση δεν ε, αρκεί. Θα πρέπει να κινηθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει αυτή η, η Ενευρυντική Επιτροπή να γίνει ένα διακυβερνητικό σώμα και όργανο. Ευχαριστώ και η Άννα Γκόμες που είναι υπόδειγμα συντομίας όταν μιλάει. Ναι, για τη CDD θέλω να μιλήσω εγώ. και για τους ε, αξιωμα... και τους υπαλλήλους ε, ελέγχονται οι τράπεζες ε, λόγω των ρυθμίσεων για, τους, για τα ανώτερα στελέχη. Ε, όπως είπε και ο κύριος Σενρία για την τον έλεγχο ε, της ε, κυρίας ε, Ντοσάντος, της θυγατέρως του Προέδρου της Αγγόλα. Ε, υπάρχει ανταγωνισμός προς τα κάτω με το διακρατικό φορολογικό ανταγωνισμό. έχουμε και αυτό το πρόγραμμα επενδυτών, οι χρήσες ε, βίζες. Αυτό δεν εννοούμε όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό φάτκα. Δεν είναι αυτό τώρα ε, αγώνας προς τα κάτω. Όλους τους διεφθαρμένους, όλους τους απαταιώνες ε, τους φέρνουμε εδώ και τους δίνουμε και χρυσή θεώρηση για να μείνουν. Ευχαριστούμε. David Coburn, συντονιστής του ECR. Κύριε Coburn, σας παρακαλώ για να ακούσουμε και τις ε, απαντήσεις. Ευχαριστώ. Δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη φοροδιαφυγή. Κανείς δεν θέλει κάτι τέτοιο ή τη διαφθορά. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την αποτελεσματική φορολόγηση. Δηλαδή το σκεπτικό ότι όλες, όλα τα κράτη είναι σωστά και δίκαια φορολογικά είναι απλά μπουρδα. Ο κόσμος προσπαθεί να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία από κυβερνήσει, διεφθαρμένες, ε, σοσιαλιστικές ή ανίκανες. Δεν κληρονομούν όλοι τον πλούτο, κάποιοι δουλεύουν σκληρά και θέλουν να τον αφήσουν στα παιδιά τους. Και γιατί όχι, δικά του είναι, αυτοί τα βγάλανε. Ο φορολογικός ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών ενθαρρύνει την αποτελεσματικότητα και την ορθή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, Αλλιώ οι κυβερνήσει θα σπαταλούν ακόμη πιο απλόχερα από ό,τι συνήθω. Δεν είναι λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις καλές και σωστές. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να προστατεύσει την περιουσία του. Μην το ξεχνάμε. Μπορεί να υπάρχει κυνήγι μαγισσών δικαίω για τους διεφθαρμένου ή του φοροφυγάδε. Και σωστά. Αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά αυτών οι οποίοι προσπαθούν να προστατευτούν. Τον αιώνα που μας πέρασε όταν δεσμεύονταν οι περιουσίες του κόσμου το 1940 το θυμάστε, ο κόσμος έχει δικαίωμα να προστατευτεί από διεφθαρμένες και άδικες κυβερνήσεις. Βεβαίως, ο συνάδελφος είναι συντονιστής του EFTD και όχι του ECR και ε, βεβαίως υπέρμαχος του Brexit και βεβαίως προετοιμάζεται για τον φορολογικό ανταγωνισμό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολλές και καλές παρεμβάσεις. Έχουμε ε, λίγα λεπτά ακόμα. Κύριε καθηγητά, ξεκινήστε εσείς, ε, κύριε Πίτ, και θα ακούσουμε και του υπόλοιπου. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομο. Ακούστηκαν πολλές ε, ερωτήσει, Ένα γενικό σχόλιο. Νομίζω πω υπάρχουν δύο ζητήματα επιτάπτως που δεν είναι ακριβώ τα ίδια. Το ένα είναι το εάν κάποιο είναι ειλικρινή στη φορολογία και πώ θα παρεμποδίσουμε το ξέπλυμα χρήματος και αν υπάρχει διαφάνεια, το θέμα της διαφάνειας. Το άλλο αφορά την φορολογική εναρμόνιση. Είναι δικό σας ε, ζήτημα το με τι σειρά θα ανοίξετε αυτά τα ζητήματα για να μην ε, ε, συσσωρευτούν πολλά και δεν γίνει τίποτα τελικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα ή τα ζητήματα της φορολογικής ειλικρινίας και της αποφυγής του ξεπλήματος χρήματος. Θεωρώ ειλικρινά ότι με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και το Παγκόσμιο Φόρουμ και τον ρόλο του ΩΣΑ έχουμε επιτύχει αρκετά. Δηλαδή έχουμε μπει, έχει μπει το νερό στα βλάκι. Ε, Βεβαίω όσοι θεωρούν ότι ε, εντάξει δεν ξέρουν αν είναι αρκετά αποτελεσματικοί αυτοί οι φορείς έχουν κάποιο δίκαιο. Η task force του ΩΣΑ είναι κάπως ε, τύπο λατρική σε σχέση με την ε, μονάδα καταπολέμησης διαφθοράς γιατί εμείς ε, μπήκαμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, δεν τσεκάρα μόνο την ομοθεσία και αυτό ισχύει πράγματι μετά το θέμα το οποίο ετέθη για την αυτορύθμιση Έχω τις προσωπικές μου επιφυλάξεις για το αν κάτι τέτοιο είναι καλή ιδέα. Στη δικιά μου τη χώρα, την Ελβετία, έχουμε πολύ εκτεταμένη αυτορύθμιση. Αφορά τράπεζες ε, και δικηγόρους ε, και ανθρώπου οι οποίοι έχουν τον ρόλο οικονομικών ενδιαμέσων. Οπότε είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Για το βασικό ζήτημα εδώ πέρα, για το κεφάλαιο της διαφάνειας. Ναι, οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ναι, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά τεχνικά υποσδήματα. Το θέμα των ενδιαμέσων επίσης. Είπα εγώ την άποψή μου για την αντιμετώπιση των δικηγόρων και εκεί πέρα κάτι πρέπει να κάνετε όταν θα συζητήσετε αυτή την οδηγία. Το ζήτημα των ΠΕΠΣ e που αναφέρθηκε από την ε, Πορτογαλία. Ναι, ξέρω, έχω δει τους λογαριασμούς Ντοσάντος ε, και βεβαίως αν κάποια στιγμή, ε, κάποια στιγμή λαμβάνει κάποιος 400 εκατομμύρια από την Σόναγκολ και τα μοιράζει στους φίλους του, ναι, πράγματι δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά οι κανόνες υπάρχουν, είναι ζήτημα εφαρμογής, δεν νομίζω ότι χρειάζονται νέοι νόμοι. Η Πορτογαλία έχει τους νόμους και το διεθνές επίπεδο επίσης. Υπήρχε επίσης το ζήτημα της ε, εθνικής ε, ελευθερίας ή μάλλον ενός ε, εθνικού περιθωρίου που αφορά όλα τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή επιτρέπουμε στα κράτη ε, μια κάποια ευχέρεια. Κάμια φορά αυτό είναι σωστό, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σταδιακά είναι ότι μπορεί να μειωθεί αυτή η ευχέρεια και να πούμε ότι το χύψη πράγμα δεν βοηθάει. Γι' αυτό εγώ ακριβώς πιστεύω στον μηχανισμό αυτών εποπτείας και μετά από τρεις-τέσσερις ε, γύρους σταδιακά να ε, εστιάσουμε. Λοιπόν, ένα άλλο υποθέμα το οποίο ετέθη είναι το ποια είναι η άποψή μου για το 25% το κατόφλι στις εταιρείε για να ταυτοποιούν ε, τους ε, πραγματικούς δικαιούχους. Είναι πολύ ψηλό, θεωρώ, έχετε δίκιο. Είναι πολύ εύκολο να έχει κάποιος ένα κατόφλι 25% και να μην φαίνεται άρα. Και μια τελευταία ερώτηση στο πλαίσιο αυτό, πολύ συγκεκριμένη, το θέμα της ε, διαδοχής των διαθήκων. Υπάρχει σε κάποιες, υπάρχουν σε κάποιες χώρες κάποιοι κανόνες ελάχιστοι για τις κληρονομιές και βεβαίως αν χρησιμοποιηθούν αυτές οι offshore, οι υπεράκτης για να παρακαμφθούν οι κανόνες είναι άδικο προφανώς. Ε, και άλλες χώρες βεβαίως δεν έχουν τέτοιους ε, κανόνες και επιτρέπεται να υπάρχει κάποιο καταπίστευμα το οποίο θα ορίζει ποιοι θα είναι οι κληρονόμοι. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε έχει απαντήσει και γραπτό στις ερωτήσεις ο καθηγητής. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Γκρότ. Ja, even eh, twee opmerkingen. was één vraag ε, Η φάκελη του Παναμά είναι πάνω από 700 υποθέσεις οι οποίες απασχολούν αυτή τη στιγμή τις ε, φορολογικές αρχές ε, και 100 με 150 από αυτές ε, πραγματικά θα έχουν συνέχεια. Οπότε υπάρχει βεβαίως και μια σχετικά υψηλή προστασία όσον αφορά τους ε, πληροφοριοδότες και θα περικοπεί και το θα περιοριστεί το επαγγελματικό απόρριτο των δικηγόρων και βεβαίως ε, υπάρχει αυτό το κατόφλι το 25% που είπατε για να ταυτοποιείται ο πραγματικός δικαιούχος. Ε, εμείς ε, όμως ε, έχουμε περάσει νόμο στην Ολλανδία ο οποίος θα αφορά όλους τους μετόχους κάτω από το 25% αδιακρίτως χωρίς κατόφλι και ελπίζουμε ε, πράγματι, ε, μάλλον έχουμε καταθέσει το νόμο και ελπίζουμε τελικά να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο να υπάρξει πλειοψηφία. Λοιπόν, σα ευχαριστώ. Κύριε Λάουι. Να απαντήσω στον Πορτογάλο συνάδελφο και στον κύριο Μπαγκή. 239 υποθέσεις τώρα περνάνε από την Ειδική Επίτροπη των ε, Φορολογικών η ICG είχε 700 ε, ε, ε, υποθέσεις επίσης και θα περιμένω το μεταποτελέσμα όσον αφορά τους ενδιάμεσους και συγκεκριμένα τις εταιρείες consulting, αυτό το Big Four, ναι, ότι κάνουν οικονομικούς ελέγχους και ταυτόχρονα δίνουν φοροτεχνικού χαρακτήρα συμβουλές. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι, θα γίνει εάν ε, το, το τμήμα που κάνει τις, ε, το, τους ελέγχους τελικά ε, θοπεύει τους πελάτες για να χορηγήσει κατόπιν τις συμβουλές. Άρα ακριβώς αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους νομοθεσία που να είναι αποτελεσματική. Ναι, θα πρέπει να έχουμε όλοι μαζί ένα κατάλογο για τους παραδείσους και θα πρέπει να έχουμε κοινέ βάσει δεδομένων πολύ σημαντικό και να έχουμε και πλήρη αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων. Μετά έχετε δίκιο. Εμείς τώρα προσπαθούμε στο Βέλγιο να έχουμε ένα καινούριο μητρό για τι εταιρείε και να μην έχουμε πλέον ε, αχύρα ανθρώπους και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν και η χώρα μα και οι του. Ο κύριος σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτά που είπε ο τελευταίος ε, συναδελφός από πλευράς ε, ε, περιεχομένου και πλευράς με σόκαρε, γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την Apple και τους υπόλοιπους με τα όσα γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που κάνει η Ιρλανδία να λέμε ότι είναι κάτι σαν ναζισμός. Ε, αυτό είναι ε, αυτό, σοκάρει να τα ακούει κανείς, ιδίως σε αυτόν εδώ το χώρο. Τέλος πάντων, αυτή η αναχώρα ε, υποβολή των αναφορών θα πρέπει να γίνεται, αλλά δεν είναι στριπτής. Είναι αυτά, αυτά τα στοιχεία, τα αριθμητικά χρειάζεται συνεργασία. Σε Γερμανία και Αυστρία είναι δημόσια αυτά τα στοιχεία και χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό το μητρό για τις εταιρείε. Δεν είναι θέμα απορρίτου επομένως. Μπορεί να υπάρχει επομένως συνεργασία και να υπάρχει και δημοσιότητα. Διαφάνεια, συνεργασία και δίκαιη φορολογία. Αυτά είναι τα οι βασικοί κανόνες. Τώρα και κάτι τελευταίο. Ακούγεται φορολογικούς παραδείσους και όλα αυτά ακούγονται σαν θετικά. Ε, δεν είναι θετικά. Θα βρούμε τα πράγματα το όνομά του Αυτά είναι σκοτεινά μέρη. Τίποτα δεν ωφελούν. Δεν έχουν σχέση με όαση και παράδεισο. Αυτά είναι κάτι σαν έλος, έλος σαν, σαν βάλτος που, που ρουφάει τα λεφτά. Κύριε Κρένα, σας ευχαριστούμε. Ε, ε, θα υπάρξουν πρακτικά ούτως ή άλλως από ολόκληρη τη συνεδρία ερωτήσεις, απαντήσεις και μπορούμε να ελέγξουμε στη συνέχεια. Εγώ δεν κατάλαβα ε, τι είπε ο κύριος Κόμπερν. Ε, Μίλαγε τόσο δυνατά στα αγγλικά που δεν ακούγα τη μετάφραση στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ α, όλους που συμμετείχατε στη συζήτηση. Δεν έχουμε χρόνο πλέον για άλλα συμπεράσματα. Θα δώσω πίσω την Προεδρία στον Πρόεδρο της ε, ΕΚΟΝ. Thank you very much ε, ε, for this very interesting first session. So we can now move uh, uh, one minute. Θα συνεχίσουμε τώρα. Αν μάλλον θα κάνουμε δύο λεπτά διακοπή και μετά, μετά θα περάσουμε στη δεύτερη σύνοδο για την Τραπεζική Ένωση, την Κεφαλαιακή Ένωση για την ενιαία αγορά για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Μην φύγετε παρακαλώ από την είναι συντομότατη διακοπή.